That has been adopted. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 είναι στη σελίδα 9, αν την ψάχνετε. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 79 και εδώ με ονομαστική πέρας ψηφοφορίας Και αυτή εγκρίνεται. Συμφεστική τρία. Ψηφίζουμε. Πέρες. Εγκρίνεται. Συμβαστική τέσσερα. Άρθρο 4. Συμβαστική 4. Ψηφίζουμε. Πέραση ψηφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Επί του άρθρου 5 ψηφίζουμε. Παρακαλώ. Εγκρίνεται Επόμενη. Συμβιβαστική 6. Επί του άρθρου 6. Ψηφίζουμε. Παρακαλώ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Επί του άρθρου 7. Έναρξη ψηφοφορίας. Yes. That has been Εγκρίνεται επίση. συμβαστική 8 επί του άρθρου 8. Ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 επί του άρθρου 9. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10. Επί του άρθρου 10. Ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 επί του άρθρου 11. Και περνάμε στην κοντ 102. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 103. Κόντε 103 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. η 12 με ονομαστική. Εγκρίνεται. Οπότε η επόμενη είναι η συμβαστική 13 Έναρξη ψηφορία για την ε, συμβαστική 13. Και εδώ εγκρίνεται. Επόμενη συμβαστική 14. 14 για το νέο 14α. Ψηφίζουμε. Συμβαστική 14 επαναλαμβάνω. Δεκατέσσερα επί του νέου άρθρου 14α. Πέρασε ψηφορίας. Εγκρίνεται. Και πάμε τώρα στην 385. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 57. Της έμπλ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Κοντ 111 και λίμπε 140 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβεστική 15. Ψηφίζουμε. Ωραία, εγκρίνεται. Οπότε, επόμενη. 488 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 489 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. Κουλτ. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, ηλεκτρονική επαλήθευση. Κουλτ 64. Λάθος μου εγκρίνεται. Λίμπε 147 υπέρ κατά αποχές αλλά και εδώ η ηλεκτρονική επαλήθευση πολύ ωραία εγκρίνεται Λίμπε 148 υπέρ κατά ε, νομίζω εγκρίνεται αλλά ηλεκτρονική επαλήθευση Απορρίπτεται. Λίμπε 149. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τέσσερα ενενήντα δύο και κατά. Υπέρ κατά. Με μισό λεπτό. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. 42, 43 και 149. Απορρίπτεται. Απορρίπτονται. Τέσσερα, νέα, τέσσερα. Και λίμπε 150. Μαζί. Ψηφίζουμε. υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 16. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφορίας. Εγκρίνεται. 505, 505 έως και έμπλ 91 μαζί. Ψηφίζουμε κατά αποχές. Εγκρίνεται. Έκον 80 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 16. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Α, με συγχωρείτε, υπάρχει τυπογραφικό λάθος εδώ. Για το άρθρο 19 μιλάμε, μέσα στο 19. Συμβιβαστική, 16 ε, λέει το εγγραφό σας, ε? Όχι, είναι 17, είναι το σωστό. Η συμβαστική 17 αφορά το άρθρο 19, γιατί 16 ήδη ψηφίσαμε. Είναι τυπογραφικό το λάθος. Η τροπολογία αφορά το άρθρο 19. Ψηφίζουμε για την 17 λοιπόν πλέον. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5-15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Να επαληθεύσουμε όμως ηλεκτρονικά. Πέρας εγκρίνεται. 516 έως και 156 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Εγκρίνεται. Κούλτ 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά λάθος μου συγγνώμη εγκρίνεται 183 έως και λίμπε 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Με συγχωρείτε, όχι έχει καταπίπτει η επόμενη, άρα αύκο 65 ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται NV65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται NV70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Yeah. NV72. Yeah, yes, all this. Yeah. So we now vote on NV... NV 72 έως και NV 86 μαζί, υπέρ. Μισό λεπτό. NV 72 έως και NV 86 μαζί, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, εγκρίνονται. NV88 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. NV89 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. NB90 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. NV91 μέρος 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. NV91 μέρος 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. NV92 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. NV93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. NV95 έως και NV99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. NV 101 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. NV 102 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. NV 103 υπέρ. Κατά. Η ηλεκτρονική επαλήθευση για την 103. εγκρίνεται. Ε, είμαστε στην συμβιβαστική 17, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. Επόμενη είναι η 575. 66 και 67 η αύκο. Α, εκεί είμαστε. 66 και 67 αύκο μαζί υπέρ. Κατά. Αποχέ Εγκρίνεται. Κόντ 126 έως και λίμπε 159 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 19. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. εγκρίνεται. Έμπλ 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 3 έως και λίμπε 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 94 υπέρ κατά Α, καταπίπτει αυτή. Συγγνώμη, λάθος μου. Έμπλ 4 έω και λίμπε 3 μαζί. Υπέρ, κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 20. Ψηφίζουμε ονομαστικά. Εγκρίνεται. Τοπολογία 79 έως και αύκο 4 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. έχουν 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Favor. Κουλτ 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Κοντ 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καλτ 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Κοντ 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δύο υπέρ κατά δεν είδα καλά τα χέρια σας και πάλι ή μάλλον ηλεκτρονικά ηλεκτρονικά τροπολογία 2 όχι δεν καταπίπτει γιατί κάποιος λέει ότι καταπίπτει ας ψηφίσουμε λοιπόν ηλεκτρονικά επί της τροπολογίας 2 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ηλεκτρονικά ελέγχουμε λοιπόν την τροπολογία 80 απορρίπτεται 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αύκο 5 υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε εκρίνεται 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται λίμπε 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται καλτ 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται κοντ 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αλλά στην ελέγξουμε Κον 5. Ελέγχουμε την Κοντ 5 ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. Οχτώντα έξι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται κοντά 6 υπέρ κατά αποχές εκρίνεται έμπλου 8 υπέρ κατά θα πρέπει να την ελέγξουμε ηλεκτρονικά εγκρίνεται Λίμπε 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 90 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 91 υπέρ. Καταπίπτει 91. Καλτ. 7. Περ. Κατά. Αποχές. Δεν είδα πολλά χέρια. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά λοιπόν. Καλτ 8 λέει ο πρώτος ελέγχουμε. Εγκρίνεται. Οίκον 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται καλπ 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έκον 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αλλά ας ελέγξουμε την έκον 6 εγκρίνεται Εκον 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Εκον 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ένβι 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται λίμπε 11 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε τη λιμπέντεκα εγκρίνεται 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 4 και αυκό 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αλλά στην ελέγξουμε την τροπολογία 98 ηλεκτρονικά. Απορρίπτεται. Έχουν 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. NV10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 100 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 102 υπέρ κατά αποχές ας την ελέγξουμε εγκρίνεται. Τροπολογία 5, αύκο 8 και τροπολογία 106 από κοινού υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, εγκρίνονται. 103 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται αλλά στην ελέγξουμε. Το πολύ 103 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Απορρίπτεται. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οίκον 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται αλλά ας την ελέγξουμε ενώ έχουμε την εικόνα 10 εγκρίνεται NV11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται λίμπε 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ελέγχουμε Ελέγχουμε την 107 ηλεκτρονικά. Εκατόν λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έκον 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αυκό 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική τροπολογία 21. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 111. Όχι, διορθώνει ο πρόεδρος. Συμβαστική τροπολογία 22 υπέρ. Α, όχι, α την κάνουμε ηλεκτρονικά. Συμβαστική τροπολογία 22. Εγκρίνεται. 112 και κόντ 10 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έγκον 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 10 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Λίβε 16 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται κάλτε 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται λίπε 18 ή μάλλον ελέγχουμε την κάλτε 10 ηλεκτρονικά 115 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 116 και κοντ 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται λίμπε 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αλλά στην ελέγξουμε τη λίμπη 19 απορρίπτεται Εκατόν δεκαεννέα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 119. Απορρίπτεται. Αύκο 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται εκατόν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Λίγο 21 λέει ο πρόεδρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται λίμπε 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έμπλ 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 123 και αύκο 16 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να τα ελέγξουμε ηλεκτρονικά εγκρίνεται έκον 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Κόντ 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. κάλτι 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αύκο 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ένβι 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έκον 17 και έμπλ 14 από κοινού υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται λίβε 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 136 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και περιλαμβάνε 136 και την 17. Πάμε στην κόντ 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται κόντ 16 και λίμπε 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται καλ 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 23 άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά It has been adopted. Λάθος. 125, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Έλεγχος για την 125. Απερίφθη. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Έλεγχος για την 132. Δεκτή. Έκανα λάθος. Λίμπε 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. ΑΦΚΟ 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Εκατόν υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Απερίφθη. Κάλτ 17 υπέρ κατά αποχές απερίφθη έλεγχος Δεκτή. Δώδεκα υπέρ κατά αποχές. Θα έλεγα απερίφθη αλλά υπάρξει έλεγχος. Απερίφθη. 139 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Εκατόν σαράντα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Έλεγχος για την 140. Δεκτή. 141 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Αυκό 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 24. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεκτή. Καλτ 20 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την Καλτ 20. Απερίφθη. Λίμπε 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 149 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Έμπλ 15 υπέρ κατά Αποχές. Απερίφθη. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την Apple 15. Απερίφθη. Αύκο 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 150 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκ... Απερίφθη. Αύκο 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Αλλά έλεγχος για την 23. Δεκτή. Λίμπε 32 υπέρ. Όχι, έχει καταπέσει. Οίκον 18 υπέρ, κατά. Δεν ψηφίσατε αρκετοί, δεν κατάλαβα. Ξαναψηφίζουμε λοιπόν τη 18 έκον. Απερίφθη. Κάλτ 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 161. Α, όχι, έχει καταπέσει. Όχι, 152 με 155 υπέρ, κατά. Λοιπόν, ηλεκτρονικός έλεγχος για τις τρεις τροπολογίες. απερίφθη με πολύ μικρή διαφορά. 161 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Έμπλ 26 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Κόντ 22 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 14 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Έμπλ 16 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Έμπλ 17 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 156 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Ένβι 13 και κόντι 23 από κοινού υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Κάλτ 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την Κάλτ 22. Απερίφθη. Έκον 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 25 Δεκτή. 159 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. απερίφθη 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Έκον 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Α, συγγνώμη. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την έκον 20. Νομίζω ότι έγινε δεκτή, αλλά έκανα λάθος. Δεκτή. Αύκο 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Έλεγχος Αύκο 24. Απερίφθη. Εκατόν Με έμπλ 18 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τις τρεις τροπολογίες. Απερίφθη. Κάλτη 25 και 26 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 165 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. ΕΝΒΙ 16 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Συμβιβαστική 26. Ψηφίζεται. Δεκτή. Περνάμε τώρα στην 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Αυκό 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 16 παρακαλώ. Απερίφθη. 167 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Κάλτ 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. κόντι 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Λίμπε 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 27. Τίθεται σε ψηφοφορία. Δεκτή. 170 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. NV22 υπέρ. Κατά. Αποχές. ΕΝΒ 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη ηλεκτρονικός έλεγχος για την M22 τελικά. Απερίφθη. Συμβιβαστή. Εκόντι 29 μάλλον. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Κάλτι 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ελέγχουμε την κόλτ 28. Απερίφθη. Εκατόν εβδομήντα ένα. Ονομαστική κλίση. Απερίφθη. 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή Κοντ 31 υπέρ κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την Κοντ 31. Δεκτή. Κόμπι 28. Ψηφίζεται. Δεκτή. του 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 174 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 175 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Καλτ 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 176 υπέρ κατά αποχές δεκτή κοντ 33 υπέρ κατά αποχές απερίφθη κοντ 34 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 177 υπέρ κατά αποχές δεκτή έκον 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Αύκο 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Κόντ 35 και Λίμπε 43 από κοινού υπέρ κατά αποχές δεκτή. 178 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Λίμπε 44 υπέρ κατά αποχές δεκτή.

Απερίφθησαν. 45 και ένβι 19 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθησαν. Συμβιβαστική 29. Ψηφίζεται. Δεκτή. Συμβιβαστική 30. Ψηφίζεται. Δεκτή. Συμβιβαστική 31. Ψηφίζεται. Δεκτή. Συμβιβαστική 32 ψηφίζεται. Δεκτή. Συμβιβαστική 33 ψηφίζεται. Δεκτή. Τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 34 υπέρ. Δεκτή. 196 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Κόντου 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Κοντ 37 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Κοντ 43 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 197. μέχρι και τη Λίμπε 52 από κοινού υπέρ κατά, αποχές, απερίθησαν 198 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. NV22 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Συμβιβαστική 35, άρχεται η ψηφοφορία. δεκτή. NV23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την nv 23 Απερίφθη. Συμβιβαστική 36 ψηφίζεται. Δεκτή. 25 και 45 κοντ. Α, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος διορθώνει. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 25. Απερίφθη. Κόντο 45 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 200 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Λίμπε 54 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 201 υπέρ κατά αποχές Απερίφθη. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 201. Απερίφθη. 202 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 202 ηλεκτρονικός έλεγχος. Δεκτή. 203 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Καλτ 38 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 37 ψηφίζεται. Δεκτή. Αυτό σημαίνει ότι πηγαίνουμε στην 206 μέχρι τη Λίμπε 55 υπέρ κατά αποχές δεκτές. Καλτ 39 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 207 υπέρ κατά αποχές δεκτή ηλεκτρονικός έλεγχος για την 207. Δεκτή. 208. Συγγνώμη, κάλτ 40 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 208 υπέρ κατά δεν μπορώ να καταλάβω τι ψηφίζετε ψηφίζουμε ηλεκτρονικά δεκτή 209 υπέρ κατά αποχές απερίφη συμβιβαστική 38 ψηφίζεται Δεκτή. Περνάμε στη συμβιβαστική 39. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεκτή. Συνεχίζουμε με την Apple 30. Όχι, έχει καταπέσει λέει η γραμματέας. Okay, okay, okay, that's right, that's right, that's right. So we are at... Λοιπόν, είμαστε τώρα στην 28. Ψηφίζουμε την 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. 29 και έκον 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτές. Λίμπε 59 υπέρ. Κατά. Λίμπε 59 επαναλαμβάνω. Ψηφίζουμε για μια ακόμη φορά υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 2-18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Καλτ 42 και Έμπλ 31 μαζί Υπερκατά αποχές δεκτή, δεκτές μάλλον. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την ΚΑΛΤ 43, 42 συγγνώμη. Απερίφθη η ΚΑΛΤ 42. ΚΑΛΤ 43 τώρα, κατά αποχές δεκτή. Το σύνολο του ψηφίσματος ηλεκτρονικά. Yep. Yes. Yeah. Mm mm-hmm. Δεκτή. Και θα πρέπει να πάρουμε και την απόφαση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Ηλεκτρονικά ψηφίζεται. Εντάξει. Λοιπόν, συγχαρητήρια στην κυρία Ροζιέχ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σύντομα θέλω να ευχαριστήσω το σύνολο των σκιωδών. Η διαπραγμάτευση είχε ένταση αλλά ήταν χρήσιμη και αυτό φαίνεται στο αποτέλεσμα. Ελπίζω να ευχαριστήσω όλους που πήραν μέρος και ελπίζω το Συμβούλιο να δεχθεί τις θέσεις μας η οποία είναι θα έλεγα χρήσιμη στην προοπτική της προστασίας αυτών που μαρτυρούν προς το δημόσιο συμφέρον. Νομίζω ότι αξίζουμε ε, διάλειμμα 5 λεπτών. Πολύ

Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν με ψηφορία. Έκθεση του κυρίου Ζιεύκα επί της χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου. Είστε έτοιμοι. Τροπολογία 103 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. that has Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2.33 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 2.34 και 2.35 μαζί υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 2, 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.47 και 2.48 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2, 7, 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 και 49 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και για την 52 ηλεκτρονικά απορρίπτεται ήταν 52 λέει ο πρόεδρος τώρα 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 έως και 62 μαζί ψηφίσουμε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 84 και 86 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 87 υπέρ. Α, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 88 υπέρ και 89 88 και 89 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 90 υπέρ κατά αποχέ. Α, να το επαληθεύσουμε καλύτερα ηλεκτρονικά γιατί είναι 90 εγκρίνεται 91 και 92 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 95 υπέρ κατά Δεν είμαι σίγουρος για την 95 ηλεκτρονικός έλεγχος. Εγκρίνεται. 96 και 97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επί του συνόλου. Τώρα ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Ζιεύκα. Και συνεχίζουμε με άλλη μια θέση του κύριου Ζιεύκα. Επιτάχυνση ρύθμισης εμπορικών διαφόρων. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά εποχές Εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. εποχές Εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. εποχές Εγκρίνεται. 28 κατά εποχές Εγκρίνεται 30 υπέρ κατά εποχές Απορρίπτεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ με συγχωρείτε καταπίπτει λέει 37 λέει ο πρόεδρος κατά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 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 57 λέει ο πρόεδρος. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για την 60 εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 65 κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 68 μάλλον αποχές απορρίπτεται 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ κατά αποχές η ηλεκτρονική επαλήθευση ε, για την 73 εγκρίνεται 75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 Απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε επί του συνόλου ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στον κύριο Σβιεφκά. Και τώρα έκθεση του κ. Ζαμίτ. Προαγωγή των θεμητών κανόνων και τη διαφάνεια για του χρήστε, του επιγραμμικούς χρήστε υπηρεσιών. Ε, συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 113, 118 μάλλον λέει πρόεδρο. Κα, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση. Νομίζω απορρίφθηκε, αλλά It has been adopted. Εγκρίνεται. 119 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 126 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ κατά να ελέγξουμε την τροπολογία 135 ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται, στο συγγνώμη. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 143 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 153 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 180 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται καταπίπτει μετά συμβαστική τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 205 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 206 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 238 υπέρ, κατά, να ελέγξουμε την τροπολογία 238 ηλεκτρονικά. Εκρίνεται. Ξέρω ότι είναι κουραστικό, αλλά πρέπει να με σιγούζετε τα χέρια. 239 υπέρ. Κατά αποχές δεν είμαι σίγουρος. Ηλεκτρονικά λοιπόν ελέγχουμε. Απορρίπτεται. 240 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 250 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 251 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 252 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 253 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 254 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ. 256 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 257. Α, όχι, 257. 258 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 259 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 260 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 281 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 317. 317 υπέρ. Κατά. Ξανά. 317. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 320 Όχι, 3.18 υπέρ. 3.18 υπέρ. the, the, the reference is incorrect. Είμαστε στην τροπολογία 318 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 320 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 321 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 323 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 324 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 325 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 19 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 326 και 327 από κοινού υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται βασική τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά να ελέγξουμε την τροπολογία 45 ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά. Πρέπει να ελέγξω και την 46 ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 85 υπέρ κατά αποχές 85 ας την ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. 86 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 87 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 88 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται Ελέγχουμε τροπολογία 88. Εγκρίνεται. 89 υπέρ. Κατά. 8 αποχές. Απορρίπτεται. 90 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 92 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε την 92 ηλεκτρονικά okay. εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 96 υπέρ κατά ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 96 εγκρίνεται συμβαστική 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 29 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 30 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 103 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 105 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 112 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και ψηφίζουμε επί του συνόλου του σχεδίου γνωμοδότησης ηλεκτρονικά. Βλέπετε λοιπόν τα συγχαρητήριά, τα συγχαρητήριά μας στον κύριο Ζάμετ. Τώρα μία έκθεση της κυρίας Κάουφμαν σε ό,τι αφορά τη θέσπιση του προγράμματος για τα δικαιώματα και για τις αξίες. Συμβαστική 53 υπέρ. Α, τροπολογία, τροπολογία όχι συμβαστική. 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε την 57 ηλεκτρονικά απορρίπτεται 61 υπέρ καταπίπτει, καταπίπτει. οπότε συμβαστική τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ κατά θα πρέπει να την ελέγξουμε την 64 ηλεκτρονικά Συμβαστική τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ, κατά, να ελέγξουμε την 71 ηλεκτρονικά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 85 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 86 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 90 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται.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 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 105 και 106 κοινέ υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 108 και 109 από κοινό υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται συμβαστική τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 114 υπέρ κατά ας ελέγξουμε την τροπολογία 114 ηλεκτρονικά απορρίπτεται 115 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 120 και 121 υπέρ κατά ας ελέγξουμε 120 και 121 απορρίπτεται 122 και 123 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 128 και 129 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται συμβαστική τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές εκρίνονται 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 136 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται βιβαστική τοπολογία 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 100 ή υπέρ κατά ε, να ελέγξουμε λοιπόν τοπολογία 100 για το σημείο ή ε εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές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 κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απορρίπτεται συγγνώμη 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 έως 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται και ψηφίσουμε από το συνόλου του σχεδίου γνωμοδότησης ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται τα συγχαρητήριά μας στην κυρία Κάουφμαν. Περνάμε στην ε, ομοδότηση της κυρίας Γκέμπχαρτ ε, σε ό,τι αφορά τη θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021 έως 2027. Συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 92 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 94 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 110 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 110. Απερίφθη. 111 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 112 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 113 υπέρ κατά αποχές δεκτή 114 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 115 υπέρ κατά αποχές δεκτή 116 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 117 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 118 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή 29 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 29 δεκτή. 30 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 129 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 129. Δεκτή. 130 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 132 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 132. Δεκτή. 35 υπέρ κατά αποχές. Δεκτή. 36 υπέρ κατά αποχές. Δεκτή. 133 υπέρ κατά Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 133. Δεκτή. 134 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 135 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 38 υπέρ κατά, αποχές, δεκτή. 39 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 1 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 2 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 3 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 41 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 42 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 43 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 44 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 5 υπέρ κατά αποχές. 49 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 50 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 50. Δεκτή. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 56 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 59 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 66 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 67 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 68 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 69 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 18 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 19 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 70 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 20 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 71 υπέρ, κατά, αποχές, Απερίφθη. Το σύνολο τώρα σε ψηφοφορία. Η πρόταση ψηφίσματος. Δεκτή. Συγχαρητήρια λοιπόν στην κυρία Γκέπχαρτ. Θα συνεχίσουμε τώρα με την έκθεση του κυρίου Χρυσόγονου. για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus. 136 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 137 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. 138 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. 139 υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το 139 παρακαλώ. δεκτό. 11 υπέρ κατά αποχές δεκτό. 140 υπέρ κατά αποχές δεκτό. 141 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 142 υπέρ κατά αποχές δεκτή 143 υπέρ κατά αποχές απερίφη 143 απερίφθη 144 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 145 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 145. Δεκτή. 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 147 υπέρ κατά αποχές δεκτή 148 υπέρ κατά αποχές δεκτή 146 υπέρ κατά αποχές δεκτή 149 υπέρ κατά α, έχει καταπέσει 149 150 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 150. 155 πενήντα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για την 155. Απερίφθη με μικρή διαφορά. 156 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 159 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 158 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 161 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 162 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 160 διακόπτει ο πρόεδρος. 164 υπέρ, κατά, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 164. δεκτή. 165 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 166 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 16 υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 166. Περνάμε τώρα στο δεύτερο τμήμα της 167. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της 167. 17 υπέρ κατά αποχές 171 υπέρ κατά αποχές δεκτή 172 υπέρ κατά αποχές δεκτή 173 υπέρ κατά αποχές Παρακαλώ οι πράσινοι και οι υπόλοιποι να σηκώνετε τα χέρια σας γιατί αλλιώς θα ελέγχουμε συνεχώς. 170. Εκατόν υπέρ, κατά, αποχές δεκτή 176 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 177 υπέρ κατά αποχές δεκτό 178 υπέρ κατά αποχές δεκτό 179 υπέρ κατά αποχές δεκτό 180 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 181 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 182 υπέρ κατά αποχές δεκτή 183 υπέρ κατά αποχές απερίφθη αλλά έλεγχος για την 183 θα υπάρξει έλεγχος Απερίφθη. 184 υπέρ κατά αποχές. Απερίφθη. 185 υπέρ κατά αποχές. Απερίφθη. 21 υπέρ κατά αποχές. Απερίφθη. 22 υπέρ κατά αποχές, απερίφθη. 186 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 187 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 188 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 189 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 190 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη 191 υπέρ κατά αποχές δεκτή 192 έχει καταπέσει 193 υπέρ κατά αποχές δεκτή 194 υπέρ κατά αποχές 194 έλεγχος. Δεκτή. 195 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Κοιτάξτε, ίσως δεν βλέπω όλα τα χέρια, δεν τα σηκώνετε. 196 υπέρ κατά αποχές 197 υπέρ ηλεκτρονικός έλεγχος δεκτή 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή 200 υπέρ κατά αποχές δεκτή 201 και 24 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος adopted um, 25 in favor 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 203 υπέρ. Συγγνώμη, λάθος. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 204 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος γιατί 204. δεκτή. 205 και 27 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Ηλεκτρονικός έλεγχος και γι' αυτό. Yes. Rejected. για μια ακόμη φορά. 206 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 209 υπέρ κατά αποχές δεκτή 211 υπέρ κατά αποχές δεκτή 212 υπέρ κατά αποχές δεκτή 213 υπέρ κατά αποχές δεκτή 214 υπέρ κατά αποχές δεκτή 215 υπέρ κατά αποχές δεκτή 216 υπέρ κατά αποχές δεκτή 217 υπέρ κατά αποχές δεκτή 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή 30 υπέρ κατά αποχές δεκτή 219 υπέρ κατά αποχές δεκτή 33 υπέρ κατά αποχές δεκτή 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή 225 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 226 υπέρ κατά αποχές δεκτή 36 υπέρ κατά αποχές δεκτή 227 υπέρ κατά αποχές δεκτή 37 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.28 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.29 υπέρ κατά αποχές δεκτή ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 2.29 Απερίφη. 38 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 39 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.30 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 2.31 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 2.32 υπέρ κατά αποχές Δεκτή. 2.33 υπέρ κατά αποχές. Δεκτή. 41 υπέρ κατά αποχές. Δεκτή. 42 υπέρ κατά αποχές. Δεκτή. 2.34 και 2.35 υπέρ κατά αποχές. Δεκτή. 2.36 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 43 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 2.37 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 2.37. Δύο Συγγνώμη, 44 υπέρ κατά, αποχές, απερίφθη. 2.39 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 2.40 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 48 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 49 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 50 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 51 υπέρ κατά αποχές δεκτή 52 υπέρ κατά αποχές δεκτή 53 υπέρ κατά αποχές δεκτή 241 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρο... απερίφθη 54 υπέρ κατά αποχές δεκτή 55 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.42 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 2.43 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 2.44 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 56 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 57 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2.45 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2.46 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 58 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 59 μάλλον υπέρ κατά αποχές δεκτή. 60, 60 ε, αποχές δεκτή. 62 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 63 υπέρ κατά αποχές δεκτή 63 ε, υπέρ κατά αποχές απερίφθη 64 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 65 υπέρ κα, κατά αποχές δεκτή 66 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 1 και 68 υπέρ κατά αποχές δεκτή 67 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2 και 70 υπέρ κατά αποχές δεκτές 69 υπέρ κατά αποχές απερίφη 71 υπέρ κατά δεκτή 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή 5 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 72 υπέρ κατά αποχές δεκτή 73 υπέρ κατά αποχές δεκτή 74 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 75 υπέρ κατά αποχές δεκτή 76 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 77 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος την 77 δεκτή. 78 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 79 υπέρ 80 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 80. Adopted ε, 81 in 81 υπέρ αποχές απορρίπτεται 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 83 Α, να επαληθεύσουμε Συγγνώμη, λάθος μου εγκρίνεται 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 90 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 91 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 99 λέει πρόεδρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 100 υπέρ κατά αποχές. Να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Για την 100. Εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 103 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση για την 9. Εγκρίνεται. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές. Άλλη μία φορά παρακαλώ. Ε, δηλαδή ηλεκτρονική επαλήθευση καλύτερα. Πολύ ωραία. Εγκρίνεται. 110. 110 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 110... 118 λέει ο πρόεδρος υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 122 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 123 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 124 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος της 10 υπέρ. Κατά. Η ηλεκτρονική επαλήθευση για το δεύτερο μέρος της 10. Εγκρίνεται. 125 και 126 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 127 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 129 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 130 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 131 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 132 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 133 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 134 υπέρ, κατά αποχές απόρριπτερα 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και επί του συνόλου της γνωμοδότησης ψηφίζουμε παρακαλώ εγκρίνεται η να συνεχίσουμε χωρίς διερμηνείς, αλλά να συνεχίσουμε με κάποιες ψηφορίες. Έχουμε την κυρία Γκέπχαρτ τώρα. Εμπόριο επί συγκεκριμένων, εμπόριο συγκεκριμένων εμπορευμάτων. Okay, Εγκρίνεται. Και έχουμε και άλλη μια γνώμη τη κυρία Γκέριγκερ. Αναδιοργάνωση Ευρωπαϊκού Δικτύου. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια στην κυρία Κέρνιγκερ και σε όλους εσάς βεβαίως.